αξία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ταυτόχρονα θα αρχίσουμε να εγείρουμε το ζήτημα αυτό με τις αρχές της Μαλαισίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Πίμπαλξ. Έξι προτάσεις ψηφισμάτων έχουν κατεθεί. Β. 7.07.09.2010 των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Β. 7.07.10.2010 7-11 ε, του 2010 των Φιλελευθέρων, 7-18 2010 των Πρασίνων και 7-27 2010 του ΕΛΚ, 7-29-2010 ε, της ΓΚΟΕ και 7-10-2010 της ΕΣΥΑΡ. Τώρα έχουμε το θέμα της ε, Ουγκάντα με τον λεγόμενο νόμο Μπαχάτη. Παρακαλώ. Κύριε Δεκεζέχ. Εδώ και ένα χρόνο ακριβώς, Πρόεδρε, συζητούσαμε στο ίδιο αυτό αμφιθέατρο ένα ψήφισμα σχετικό με, τον νόμο Μπαχάτη και τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και των λεσβιών. Γιατί ξαναρχόμαστε ένα χρόνο μετά με ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Διότι ακριβώς δεν έχει λήξει το πρόβλημα. Το εμβαγγελικό κείμνημα The Family, η οικογένεια που υποκίνησε αυτό το νόμο Μπαχάντη φαίνεται ότι δεν υποχωρεί και βλέπουμε ότι επανέρχεται με μεγαλύτερη έμφαση και ένταση αυτός ο νόμος στην Ουγκάντα. Ο δεύτερος λόγος είναι τον Οκτώβριο και Νοέμβριο που μας πέρασαν το περιοδικό Rolling Stone της Ουγκάντας ε, έκανε αυτό που ονομάζεται naming and shaming, δηλαδή κατήγγειλε δημόσια με, τα ονόματά τους ε, ομοφιλοφίλους της Ουγκάντας οι οποίοι διώχθηκαν, εκδιώ, ε, διώχθηκαν, ε, προπυλακίστηκαν, ακόμη και βιάστηκαν και τώρα κρύβονται για να σωθούν. Έχει δηλαδή ξεκινήσει ένα πραγματικό ανθρωποκυνηγητό στην Ουγγάντα. Εν τω μεταξύ 13 μονοκράτη της Αφρικής αναγνωρίζουν δικαιώματα για τους ομοφιλοφίλους. Τα υπόλοιπα κράτη έχουν πολύ διαφορετικές και αποκλίνουσες νομοθεσίες, αλλά υπάρχουν κράτη τα οποία ε, απειλούν ακόμη με θάνατο την ομοφιλοφιλία, όπως η Μαυρετανία, το Σουδάν και η Βόρεια Νιγηρία. Υπάρχουν κάποια κράτη λοιπόν από την ΑΚΕΟ που όταν συνομιλούμε για τα προβλήματα των ομοφιλοφίλων μας λένε ναι καταλαβαίνουμε μας ενοχλούν αυτά τα θέματα και όλοι μας, εν... μας παρενοχλούν για τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων αφήστε μας γιατί είναι η ιδιαιτερότητά μας πολιτιστική. Η δε δική μας απάντηση είναι όχι πρόκειται για πολιτιστικές, για, πρόκειται για οικουμενικές αξίες δεν μπορούν να... Ευχαριστώ κύριε Ντεκάιζερ. Για ένα λεπτό κύριος ε, Τάνοκ. Στην Αφρική τα ήθη είναι πολύ συντηρητικά. Σε πολλές χώρες της Αφρικής δυστυχώς απαγορεύεται ομοφιλοφιλία. Και είναι πολύ δύσκολο να προωθηθούν τα θέματα ίσων δικαιωμάτων για τους ομοφιλοφίλους. Στη Δύση θεωρούμε ότι αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα, ενώ οι Αφρικανοί πιστεύουν ότι προσπαθούν να περάσουν τις πιο, τα πιο χαλαρά δυτικά ήθη στις αφρικανικές ε, κοινωνίες που έχουν άλλα ήθη και έθιμα. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν να δικαιολογήσει την ομοφιλοφιλή ομοφιλοφοβία που υπάρχει σε πολλές χώρες Αφρικής και τροφοδοτείται ακόμα και από κυβερνήσει. Η Ουγγάντα είναι ένα από τα κράτη τα οποία χαρακτηρίζονται για αυτή την ιστερία. Υποστηρίζουν ένα νόμο ο οποίο ε, εφαρμόζει θανατική ποινή ή και στην καλύτερη περίπτωση ισόβια δεσμά στους ομοφιλόφιλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το απορρίπτω μεταβδελιγμίας γιατί είναι μια πραγματική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ουγγάντα είναι μια χώρα όπου η πλειοψηφία των ανθρώπων ζουν μονάχα με ένα δολάριο το χρόνο. Ίσως οι νομοθέτες της χώρας αυτής μπορούν να βρουν καλύτερου τρόπους να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τη ε, χώρα αυτή από το να κυνηγούν του ομοφυλόφιλου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Ακολουθεί για ένα λεπτό η κυρία Σάκη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία... κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Ο νόμος κατά των ομοφιλοφίλων στην ε, Ουγκάντα προβλέπει φυλάκιση από 7 χρόνια ως ισόβια δεσμά, ακόμα και θανατική ποινή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταδικάσει εκπεφρασμένα αυτή την νομοθεσία. Δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε ευρωπαϊκά πρότυπα σε άλλους, αλλά δεν μπορεί να αποσύσει έτσι την ευθύνη η Ουγκάντα που έχει να προστατέψει τους πολίτες της και να την χάνουν επιθέσει οι πολίτες τους επί τη βάση σεξουαλικού προσανατολισμού. Οι απειλές και το κλίμα ε, φόβου φάνηκε από την τοπική εφημερίδα Rolling Stone, η οποία δημοσίευσε στον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ονόματα ανθρώπων που θεωρούνται ότι ήταν ομοφιλόφιλοι, ζητώντας από τους αναγνώστες του να τους επιτεθούν. Πολλά άτομα πράγματι έτυχαν επιθέσεω. Πολύ η ομοφιλοφίλια είναι ε, νόμιμη μόνο σε 13 αφρικανικά κράτη και είναι ποινικό αδίκημα σε άλλα 38 στο Σουδάν και τη Βόρεια Νιγηρία τιμωρείται με θάνατο. Οι αρχές του Ουγγάντας πρέπει να συμμορφωθούν με τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με την ε, Συμφωνία της Κοτονού και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η... όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνουν την απαραίτητη προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι όλοι απολαμβάνουν των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σάκη. Ακολουθεί για μισή λεπτό ο κύριος Ρωμέβα και Ρουέδα. ο νόμος Μαχάτη στο Ουγανδικό Κοινοβούλιο που προβλέπει την ε, κόλαση των ομοφιλοφιλοκών πράξεων με ποινές από 7 ε, χρόνια κάθριξη έως θανατική ποινή είναι, ανα... είναι απαράδεκτη. Μόνο σε 13 χώρες όπως αναφέρθηκε είναι νόμιμη ομοφιλοφιλία και σε 38 χώρες είναι ποινικό αδίκημα. Στη Μαυριτανία, το Σουδάν και στη Βόρεια Νιγηρία η τιμωρία είναι ο θάνατος. Γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε και πάλι ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι μέσα στα ατομικά δικαιώματα ιδιωτικότητος, υποστηρίζεται από το Παγκόσμιο Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσα στο οποίο αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία έκφρασης και επίσης προστασία σεξουαλικού προσανατολισμού. Γι' αυτό θέλουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια αναμόκλευσης των παθών και του μίσους εναντίον των ε, ατόμων που δεν έχουν την κυρίαρχη σεξουαλική προτίμηση. Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι παράνομη αυτή η νομοθεσία σύμφωνα με την Συμφωνία της Κοτονού. Πρέπει λοιπόν οι αρχές της, ε, ε, του Συμβουλίου ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να τονίσουν τη σημασία να υπάρχει πλήρης απολαβή δικαιωμάτων από τις λεσβείες, τους ομοφιλόφιλους, τους αμφίφιλους και τους ε, ε μετασεξουαλικούς. Ένα λεπτό κύριο Κάτσμαρέκ. Διεμφυλικούς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, οι διακρίσεις οι σχετικές ε, με τον γενετήσιο προσανατολισμό ε, στην Ουγκάντα θα πρέπει να καταργηθούν. Την Ουγκάντα δυστυχώς ε, την στηρίζουν κάποιες αφρικανικές χώρες οι οποίες δεν δέχονται τις πιέσεις που ασκεί η, δυτική, διεθνής κοινότητα και τα δυτικά κράτη ιδιαίτερως. Εδώ έχουμε να κάνουμε όμως με ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αμφισβητούν στην πλειονότητά τους τα αφρικανικά κράτη. Και έτσι μιλούμε εμείς για βασικές ανθρώπινες αξίες, αλλά ισόταμοι ακουόντων, γιατί εκείνοι μας λένε «Α, ε, πρόκειται για ιδιαιτερότητα δική μας». Πρέπει λοιπόν να απαγορευθούν αυτοί οι νόμοι, πρέπει να αντισταθούμε εμείς και να ασκηθεί στο βαθμό του δυνατού η πίεση ώστε να μην περάσουν. Ευχαριστώ πολύ για δύο λεπτά κυρία Βεργιά. Η Ουγγάντα όντως συγκαταλέγεται μεταξύ των αφρικανικών κρατών που ε, τιμωρούν βαρύτατα την ομοφιλοφιλία και μάλιστα έχει και μια από τις πιο σκληρές διότι υπό τον έλεγχο των Ευαγγελικών Αμερικανών Ιεραπαστόλων έχει ξεκινήσει με τον ε, βουλευτή Μπαχάτη ε, ένα ανθρωποκυνηγητό εις βάρος των ομοφιλοφίλων. Μουσουλμάνοι λοιπόν και χριστιανοί και πρόκειται για μια πρώτη εκδήλωση συνεργασίας τέτοια στην ε, χώρα αυτήν αντέδρασαν για να αντισταθούν σε αυτόν τον νόμο και ένας χριστιανός ευαγγελικός ιερέας, ο οποίος στάχθηκε με το πλευρό των ομοφυλοφύλων και αγωνίστηκε για τα δικαιώματά τους, ε, αποσχηματοποιήθηκε. Κινδυνεύουν λοιπόν με την ποινή του θανάτου οι ομοφιλόφιλοι εάν υπάρχει υπόνοια συνέβρεσης με ανηλίκους ή ε, ιού του HIV-AIDS. Το δε περιοδικό Rolling Stone τη Ουγγάνδας που δεν έχει καμία σχέση με το, αμερικανικό πολυγνω... αγγλικό που γνωρίζουμε έχει δημοσιεύσει ονόματα ε, ομοφιλοφίλων με τίτλο πηχαίο «Κρεμάστε τους». Και ναι, μεν απαγορεύτηκε, αλλά ήταν πια πολύ αργά, γιατί όπως υπόθηκε υπέστησαν πολλά δεινά αυτοί οι άνθρωποι. Έχει αντιμετωπιστεί ως ε, μία μάστιγα που εισήχθη από την Ευρώπη ομοφιλοφιλία. Θεωρείται δηλαδή ότι οι Ευρωπαίοι την έφεραν στην Αφρικανική αυτή χώρα για να καταρακώσουν το αιωσύστημα της ηθικής, της κοινωνικής ηθικής. Νομίζω ότι θα πρέπει να το στηρίξουμε και πάνω απ' όλα να βοηθήσουμε όσους ε, ομοφιλοφίλους της Ουκάνδας υφίστανται αυτές τις διώξεις, όπως κάνουμε για κάθε θύμα βασανιστήριων και πάθαπης μεταχείρισης. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Τώρα, κύριε Μακοβέη πρώτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με ανησυχεί βαθύτατα η ε, εισαγωγή νομοθετήματος το οποίο απαγορεύει τη συνέβρεση μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου σε ιδιωτικό χώρο. Φαίνεται ότι προχωρεί αυτή η νομοθεσία και ενώ ήδη υπήρχε μια σχετική απαγόρευση, ο νόμος Μπαχάτη επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τα ε, πράγματα. Με τη νέα νομοθεσία θα ενταθεί το κλίμα του φόβου και της μυσαλλοδοξίας σε μια περιοχή όπου ήδη επικρατεί ε, αδιακρισία ως προς τον ιδιωτικό βίο των ανθρώπων και κινδυνεύει η ζωή των ομοφιλοφίλων. Στην Ουγγάντα δεν θα έχει κανένα νόημα ο όρος ανθρώπινη αξιοπρέπεια αν εισαχθεί αυτή η νομοθεσία και δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μακοβέη. Ο επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό είναι ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά, πολλά έχουν αλλάξει το τελευταίο χρόνο. Στις 23 Νοεμβρίου το Κοινοβούλιο μας τόνισε τη σημασία της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μη διάκρισης μέσα στα πλαίσια και της εταιρική μας σχέση με την ε, ε, σχέση μας με τις χώρες ΑΚΕ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις όταν υπάρχει έλλειψη σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των άλλων όταν πρόκειται για διακρίσεις οι οποίες βασίζονται σε σεξουαλικό προσανατολισμό. Η διαφορά είναι ότι αυτές οι χώρες διαλέγουν να λειτουργούν μαζί μας, θέλουν να έχουν μια εταιρική σχέση. Έχουμε τη συμφωνία με τις χώρες αυτές, έχουμε τις συμφωνίες Κοτονού, ω εκ τούτου ζητούμε από αυτές τις χώρες να συμμετάσχουν σε συνεργασία μαζί μας επί τη βάση κοινών ε, οικουμενικών αρχών που δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Εάν δεν το θέλουν, ζητώ από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να αναλάβουν τις απαραίτητες κυρώσεις για να τονίσουν το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τι αξίες τις οποίες θα προασπίσει. Και το μέλλον της στρατηγικής σχέσης μας με την Αφρική εξαρτάται από το ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες δράσεις βάσει της εταιρικής σχέσης χωρίς καμία μορφή διάκρισης μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η σεξουαλική προτίμηση. Δεν πρόκειται, έχω ένα 1,5 λεπτό κύριε Πρόεδρε, δεν είναι θέμα απεικιοκρατία το να υποστηρίζει κανεί τα δικαιώματα των άλλων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι αδιέρετα και οικουμενικά. Το να κοιτάμε αδιάφορα αλλού όταν υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό είναι μία μορφή συνενοχή. Δεν μπορεί κανεί να παροτρύνει την ομοφιλοφιλία. Δεν μπορεί κανείς που έχει σώστας φρένας να πει σήμερα θα δεχτώ ότι είμαι ομοφιλόφιλος. Θα τον καταδώσουν οι γείτονέ του στην αστυνομία, θα καταλήξει στη φυλακή. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε αυτά τα δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Πράγματι, ήταν ένα μισή λεπτό ο χρόνος σας. Η κυρία Τάιν, ένα λεπτό μόναχα. Κύριε Πρόεδρε η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Χάρτα του Συμβουλίου τη Ευρώπη απαγορεύουν τη διάξηση τη βάση σεξουαλικού προσανατολισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο έχει υποχρεώσει το δικό τη έδαφο, τη δική τη επικράτεια σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει επίση και ευθύνη βάσει των συμφωνιών τη με τρίτε χώρε να εξασφαλίσει την τήρηση αυτών των δικαιωμάτων. Η Ουγγάντα έχει μια σχέση συν, και λαμβάνει χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παραβιάσουν ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ορθώσει τη φωνή τη όταν γίνονται τέτοιου είδου παραβιάσει. Πρέπει να τηρηθεί η Συμφωνία Κοτονού, την οποία έχουν υπογράψει ελευθέρω χώρε όπω η Ουγγάντα και αυτή είναι το πλαίσιο συνεργασία μα με τι χώρε ΑΚΕ. Έχουμε ζητήσει πριν από δύο χρόνια ζητήσει από την Ουγγάντα να μην προχωρήσει στο νομοθέτημα αυτό και την ποινικοποίηση των ομοφιλοφιλών. Ενδεχομένως η κατάσταση έχει χειροτερέψει, έχουμε μακρύτερες ποινές φυλάκισης, ακόμα και κίνδυνο θανατικής ποινής. Ε, δεν έχουν καρποφορήσει προσπάθειες να αντιταχθούν οι διαδηλωτέ και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι σε αυτού του νόμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει όμω να παρέμβει σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τάινα, ακολουθεί ο κύριο Τσαρνέτσκι για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική η συζήτηση. Η Ουγκάντα δεν είναι μεμονωμένη στην επιβολή διακρίσεων στα θέματα αυτά. Τα τρία τέταρτα, αν δεν απατώ, με των κρατών της Αφρικής έχουν πολύ αυστηρές νομοθετικές διατάξεις νομοθεσίε για τα θέματα αυτά και εν γέννη επιβάλλουν διακριτική μεταχείριση. Το πρόβλημα δεν αφορά δηλαδή μόνο την Ουγγάντα αλλά ολόκληρη την Ήπειρο και ολόκληρη την αφρικανική κουλτούρα, λέει ο μιλητής. Δεύτερον, η Ουγγάντα δεν είναι πρωτοπόρος στην προστασία των δικαιωμάτων στην Αφρική. Εδώ πρόκειται για ένα ίσον ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έστω ας το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λέω πρόεδρος, ο κ. Μάιερ δυστυχώς δεν είναι παρόν. Προχωρώ λοιπόν στον κατάλογο των ομιλητών η κυρία Κρέτσου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το ψήφισμά μα ασχολείται με βαρύτατε ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώ στην Αφρική η ομοφιλοφιλία αποτελεί κολάσιμο αδίκημα. Από τα 38, 38 ε, είναι τα κράτη της Αφρικής τα οποία επιβάλλουν ποινικέ κυρώσεις για την ομοφιλοφιλία και μόνο σε 13 είναι νόμιμοι. Εδώ με ποινές που φτάνουν μέχρι και το θάνατο έχουμε να κάνουμε με κατάφορες των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Γι' αυτό ήρθε η ώρα πλέον να καταγγείλουμε την ε, κατάσταση αυτή πριν να ε, πληγούν και άλλοι άνθρωποι όπως αυτοί που καταγγέλθηκαν από το περιοδικό Rolling Stone. Η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι βασικό στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει αποφασιστικά να δράσουν και μέσα από τις διεθνείς του συμφωνίες να επιβάλλουν την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και από την Ουγγάντα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρετσού. Ίσα ίσα προλάβατε το χρόνο και τώρα περάμε στη διαδικασία Κατστιάη. Ο κύριος Πρέντα έχει στήσει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν το θέμα της ομοφιλοφιλίας στην Ουγγάντα πριν από λίγους μήνες. Έκτοτε η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά. Πολλέ φορέ λέμε ότι η έλλειψη ειδήσεων είναι θετικά νέα. Σε αυτή την περίπτωση όμω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εάν, εάν δεν είχε εγκριθεί ο νόμο Μπαχάτη, ο νόμο Μπαχάτη δεν έχει αποσύρθει ακόμα. Είναι παρκαρισμένο στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων τη Ουγγάντα του Κοινοβουλίου τη Ουγγάντα και παρά τι προπιέσεις που ασκήθηκαν δεν έχει αποσυρθεί αυτό το νομοθέτημα. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό είναι η αντιμετώπιση των ομοφιλοφίλων με συγκροτημένη εκστρατεία που γίνεται σήμερα στην Ελπίζ, ελπίζουμε ότι οι αρχές Ουγγάντα θα δείξουν σοφροσύνη και θα τηρήσουν την αρχή τη μη διάξης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέντα για το τέλος της διαδικασίας Catch ο κύριος Χίγκινς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εκστρατεία μίσου στην Ουγγάντα εναντίον των ε, ε, ομοφιλοφίλων και λεσβιών είναι πραγματικά αποτρόπαια. Είναι μια εκστρατεία η οποία είναι καθαρά ομοφιλοφοβική που ανακοινείται από τα μέσα ενημέρωσης θέλουν να σκοτώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν εχθρούς τους και πάρα πολλοί ομοφιλόφιλοι και λεσβείες ζουν σε κατάσταση μεγάλου φόβου και ανησυχία στην ε, Ουγγάντα. Προτείνονται ακόμα και οι δημόσιες εκτελέσει αυτών των ανθρώπων. Εγώ χαιρετώ το θάρρο των μελών της ε, κοινότητας των ομοφιλοφίλων στην Ουγγάντα που κάθε μέρα αγωνίζονται εναντίον αυτού του κινδύνου για την ταυτότητά του, ακόμα και για την ζωή του. Η ομοφοβική αυτή εκστρατεία τροφοδοτείται από στρεβλώσει και ψέματα για το τι σημαίνει να είναι κανείς ομοφιλόφιλος. Το πιο ισχυρό μήνυμα θα πρέπει να πάει προς την κυβέρνηση της Ουγγάντα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ενεργή αλληλεγγύη με όλου του φορεί στην Ουγγάντα, οι οποίοι αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Θα πρέπει να του βοηθήσουμε σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη μάχη για τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το δικαίωμα να είναι κανεί αυτό το οποίο είναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χίγγινς. Για να κλείσει η συζήτηση, δίνω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Πίμπαλξ, εξ Κομισιόν. Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι. Το σχέδιο νόμου κατά των ομοφιλοφίλων που εισήχθη στο Κοινοβούλιο της Ουγκάντα ε, εγείρει πολλά ζητήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα δικαιώματα των ε, λεσβιών, ομοφιλοφίλων, διεμφυλικών και αμφιλοφίλων. Είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμερίζομαι πλήρω τι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση στην Ουγκάντα, καθώ και σε άλλε χώρε όπου κυρωτική και ε, διακριτική μεταχείριση επιβάλλεται από την νομοθεσία εις βάρος αυτών των ομάδων πολιτών. Η ποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας, όπως προβλέπεται στο σχέδιο του νόμου, παραβιάζει και βασικές υποχρεώσεις υπό τη Σύμβαση των Κοινών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, την οποία έχει προσπογράψει και η ΟΓΚΑΝΤΑ Και επίσης την διακηρυκή 6 των Ηνωμένων Εθνών για τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα των φίλων. Ετέθη το ζήτημα αυτό στην κυβέρνηση του Γκάντα σε αρκετέ περιπτώσει επικοινωνία μα και σε συνεδριάσει με τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό των Εξωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνη, είτε σε ε, συνεδριάσει τυπικού ε, διαλόγου, είτε σε επαφή με την ε, Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ουγκάντα η κυκλοφορία του περιοδικού στις 2 Οκτωβρίου του 2010 του Rolling Stone, το οποίο έδινε φωτογραφίες, ονόματα και διευθύνσεις ανθρώπων που χαρακτηρίζουν φιλόφιλους και με τίτλο «Κρεμάστε τους» ήταν μια αποτρόπαιη πράξη. Έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Την καταδικάζουμε. Η Αντιπροσωπεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ μαζί με την αντιπροσωπεία των, με τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών που είναι παρόντα στην Ουγγάντα, αλλά και με χώρε εταίρου όπω Νορβηγία, Ηνωμένε Πολιτείε, με, την, ε, με το γραφείο εκεί του είπα του εκπροσώπου τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ και μέσω τη ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ομάδα εργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αποτελεί και το επίσημο κέντρο ε, διαλόγου για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την ανάληψη δράσεω για θέματα παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ουγγάντα. Παρακολουθούμε λοιπόν την κατάσταση και διαρκώ εγείρουμε τι ανησυχίε, εκφράζουμε τι ανησυχίε μα για το σχετικό αυτό νομοθέτημα, αλλά και για άλλε δραστηριότητε ε, δίωξη των ε, ομοφιλοφίλων λεσβιών, αμφιφιλικών και αμφιφιλικών και διεμφυλικών στην Ουγγάντα Και στηρίζουμε τι οργανώσει των πολιτικών δικαιωμάτων στι προσπάθειέ του να αλλάξουν οτροπίε στου πολίτε τη χώρα, αλλά και να βελτιώσουν την κατάσταση για του ομοφυλόφιλου, λεσβείε, διεμφυλικού και επιφυλόφιλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έξι προτάσεις ψηφίσματος έχουν κατατεθεί και θα γίνει η ψηφοφορία στο τέλος της συζητήσεως. Και τώρα έχουμε τους